πολιτών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο αντιδρά στις πρωτοβουλίες των Ευρωπαίων πολιτών για να απαγορευτεί η γλυφοσάτη και να προστατευτεί ο κόσμος από τις τεξικές ουσίες. Εμείς ζητάμε ένα πιο ανεξάρτητο σύστημα με διαφάνεια. Ζητάμε έγκαιρη προειδοποίηση του κοινού από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων. Έτσι θα αυξηθεί ο έλεγχος στην αδειοδότηση ουσιών που καταναλώνουμε είτε μιλάμε για γενετικά τροποιημένα τρόφιμα, είτε για αρωματικές ουσίες, είτε για οτιδήποτε. άλλο. χάρη στους κανόνες για την έγκαιρη αποκάλυψη πληροφοριών, η ΕΦΣΑ ανοίγει τις πόρτες της στους πολίτες ε, για τα δεδομένα τα οποία παρέχει η βιομηχανία. Οποιαδήποτε πληροφορία η οποία αφορά την ασφάλεια θα αποκαλύπτεται πάντα στο κοινό. Στόχος μας λοιπόν ήταν να σταματήσουν οι πρακτικές αυτές που αφορούν την απόκρυψη δεδομένων ή μελετών που δεν ήταν ευνοϊκές και τα καταφέραμε. Δεν θέλουμε άλλη γλυφοσάτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θέλουμε άλλες αποφάσεις και κλεισμένων των θυρών και όχι άλλο τζόγο με την υγεία των ανθρώπων. Σε δύο... Σε μια ε, εποχή όπου η κινητήριος δύναμη είναι το χρήμα, η διασφάλιση των πολιτών είναι ένα σύστημα εύρωστο το οποίο θα αντέχει στις εξωτερικές πίεσεις. Χαίρομαι για το ότι η ομάδα μας απέδειξε ότι η υγεία και τα δικαιώματα είναι πάνω από τα εμπορικά συμφέροντα. Σας ευχαριστώ. Τον λόγο έχει η κυρία Χάζα Κάμπια την Κούε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εδώ και δεκαετίες επιχειρήσεις όπως η Bayer, Monsanto και συντζέντα δείχνουν, ε, ρίχνουν διαφορές ουσίες μέσω των ε, λιπασμάτων που καταλήγουν στα χωράφια και από εκεί στα τρόφιμά μας. Βλέπουμε τις καταστροφικές συνέπειες. Ε, πεθαίνουν οι μέλισσες, μειώνεται η βιοπικιλότητα, ρηπαίνεται το νερό και τα ύδατα. Τεράστιες ζημιές για ανθρώπους και ζώα. Και έρχονται τώρα εδώ πέρα και θέλουν να ξεφύγουν χάρη στην χαλαρή νομοθεσία της σύγκρουσης συμφερόντων στην ΕΦΣΑ και διαδικασίες οι οποίες βασίζονται σε προεγκεκριμένες ε, μελέτες τις οποίες έχει παραγγείλει η βιομηχανία. Ήδη χτες δόθηκε αδειοδότηση σε 30 νέα ζυζανιοκτώνα χωρίς αξιολόγηση. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Πότε θα δράσετε ως Κομισιόν αντί να ασχοληθείτε επιτέλους με την υγεία των ανθρώπων και όχι με τις μετοχές της Μπάγκερ και της Συντζέντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ε, ευχαριστώ. Τον λόγο έχει ο κύριος Χόισλινγκ. Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα είναι μια θετική μέρα για την Ευρώπη, γιατί έχουμε την ευκαιρία να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στην διαδικασία αδειοδότησης, η οποία χάθηκε με την γλυφοσάτη. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω 1,3 εκατομμύρια πολίτες που υπέγραψαν για μία πρωτοβουλία πολιτών ονόματι «Σταματήστε την γλυφοσάτη» έτσι ώστε να υπάρξει μια διαφάνεια στην διαδικασία αδειοδότησης των χημικών ουσιών στην Ευρώπη. Και γνωρίζουμε ότι το θέμα της γλυφοσάτης δεν έχει τελειώσει. Ήταν η αρχή γιατί η γλυφοσάτη εξακολουθεί να είναι αντικειμενοκριτικής και βλέπουμε ειδικά στις ΗΠΑ πως οι επιφυλάξεις είναι πάρα πολύ σοβαρές και θα δούμε το τι θα γίνει με την ε, διαδικασία αδειοδότησης. Λοιπόν, τι καταφέραμε. Υπάρχει πρόσβαση σε όλες τις μελέτες, ο καθένας μπορεί να τις διαβάσει. Όλες οι μελέτες πρέπει να δημοσιεύονται και αυτές που δεν συμφέρουν τις επιχειρήσεις και αυτά θα τα ελέγχει η ΕΦΣΑ. Ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός. Προς το συμφέρον των πολιτών και του περιβάλλοντος και όχι των επιχειρήσεων. Αυτά λοιπόν και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Και για το ΕΛΚ η κυρία Πιετικά είναι να έχει τον λόγο. Η καινοτομία και το θέμα των εμπορικών μυστικών αυτά ποτέ δεν μπορεί να προηγούνται της δημόσιας υγείας. Γι' αυτό αυτή η συμφωνία η συμφωνία όσον αφορά τη διαφάνεια της έρευνας για τα τρόφιμα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όσο πιο περίπλοκο είναι το σύστημα των τροφίμων, τόσο περισσότερες πληροφορίες έχουμε για διάφορα συστατικά. Συστατικά όπως είναι χημικά, χημικές ουσίες, νανοπλαστικά κλπ. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε όλο και ευρύτερο πεδίο έρευνας και δημοσίευση των ερευνών και αξιολόγηση του τι θεωρούμε ότι είναι ασφαλές τρόφιμο. Αυτό έχει σχεδιαστεί να κάνει η νομοθεσία. Και η περίπτωση της γλυφοσάτης οδήγησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνουν κάτι και να προχωρήσουν νέες πληροφορίες συγκρουόταν με τα συμφέροντα της δημόσιας υγείας και παρέμειναν εμπιστευτικές αυτές οι πληροφορίες. Τώρα διορθώθηκαν τα πράγματα. Το επόμενο βήμα είναι το πώς η ΕΦΣΑ θα απαιτείται να χρησιμοποιεί την αρχή της πρόληψης καλύτερα από ό,τι πριν, όταν θα δίνει εντολή για μελέτες. Ευχαριστώ πολύ. Ε, επόμενος, Μπουσόη, συνάδελφε Μπουσόη εκ μέρου του ΕΛΚ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έξοχη η πρότασή τη και ευχαριστώ και την κυρία Πιλάρα Γιούσο για την πληρέστατη έκθεσή τη. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι σημαντικότατο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να ξαναποκτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και να μεγιστοποιήσει τη διαφάνεια των επιστημονικών μελετών στον τομέα τη ασφαλεία των τροφίμων, κυρίω μετά από τι πασίγνωστα προβλήματα που αφορούν την αδειοδότηση κάποιων ευαίσθητων προϊόντων, όπω γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί ή κάποιες ενεργές ουσίες, όπως είναι νεκοτινοειδή και η ήδη διαβόητη γλυφοσάτη. Στον τριμερή διάλογο το Κοινοβούλιο πέτυχε ισορραπία, επέτυχε μια προσωρινή συμφωνία από το Συμβούλιο και καταρτίζεται μια διαδικασία αξιολόγησης που είναι ανεξάρτητη, διαφανής και συμπραβάνει όλα τα στοιχεία και θα πρέπει ε, κατευθείαν να δημοσιεύονται όλε οι μελέτε τη Υπηρεσία Τροφίμων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να υπάρχει διάλογο με την κοινωνία των πολιτών, τόσο να εξασφαλίζεται η επικράτηση του δημόσιου συμφέροντος. Όμως, για να εξασφαλιστεί η πλήρης επιτυχία του νομοθετικού πλαισίου είναι ύψη τη σημασία και δράτωμα τη ευκαιρία να απευθύνω έκκληση προ τη μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών, είναι ύψη σημασία να ενθαρρύνουν του εμπειρογνώμονε να γίνουν μέλη των ομάδων επιστημονική εξολόγηση των κινδύνων. Για... Διότι μέχρι τώρα μόνο έξι χώρε δίνουν τα δύο τρίτα του συνολικού αριθμού των εμπειρογνωμών. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ξεκινάμε τη διαδικασία Catch the Eye. Καταρχάς, κύριε Σόιντροβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στο προηγούμενο θέμα ασχοληθήκαμε με την διπλή ποιότητα των προϊόντων. Τώρα πάλι μιλούμε για την ποιότητα των προϊόντων, αλλά για την ασφάλεια των τροφίμων. Θεωρώ ότι αυτό το σημείο είναι εξίσου σημαντικό όσο το προηγούμενο με τη διπλή ποιότητα των προϊόντων. Στη συγκεκριμένη έκθεση μιλούμε για τη διαδικασία διοδότησης που θα πρέπει να στηρίζεται σε ξεκάθαρες επιστημονικές αποδείξεις και γνωματεύσεις. Θα θέλουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία που θα ενισχύσει τη διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης του κινδύνου που πραγματοποιεί ο Οργανισμός Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα θα πρέπει να απειλούμε με την πρόταση αυτή την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Θέλουμε ενισχυμένη ε, διαφάνεια για να καταρρύψουμε κάποιες θεωρίες περί συνωμοσία και να εξασφαλίσουμε σωστή πληροφόρηση και να εξασφαλίσουμε και υψηλή ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων. Αλλά να μην ξεχνούμε και την ανάγκη να σεβαστούμε το εμπορικό ε, ή βιομηχανικό απόρριτο. Η ΕΦΣΑ πιστεύω ότι θα σέβεται καλύτερα, θα εφαρμόσει καλύτερα τι διαδικασίες. Ο κ. Μαριάς. Η αξιολόγηση κινδύνου στην αλυσίδα των τροφίμων είναι κάτι σημαντικό γιατί πραγματικά υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία των καταναλωτών και νομίζω ότι πρέπει εδώ να είμαστε αποφασιστικοί. το βασικό στοιχείο είναι η ετικετοποίηση να γνωρίζουμε πραγματικά τι περιέχουν τα τρόφιμα. το δεύτερο είναι να προσέξουμε κυρία κατάινεν τις εισαγωγές από τρίτες χώρες γιατί εκεί δεν τηρούν τις προϋποθέσεις. παράδειγμα στην τουρκία καλλιεργούνται ντομάτες και άλλα αγροτικά προϊόντα με λιπάσματα τα οποία απαγορεύεται να κυκλοφορήσουν στην ίδια την ευρωπαϊκή ένωση. τρίτη περίπτωση παράνομες ελληνοποιήσεις προϊόντων δηλαδή εμφανίζονται προϊόντα ως δήθεν ελληνικά ενώ αυτό απαγορεύεται το έχω καταγγείλει επανειλημμένα παράνομη ελληνοποίηση γάλακτος που εισάγεται μέσω αλβανίας παράνομη ελληνοποίηση κρεάτων που εισάγονται μέσω σκοπίων. τα θέματα αυτά είναι σημαντικά και για την προστασία του καταναλωτή και φυσικά για το χτύπημα της απάτης και επιπλέον για την προστασία και σε επίπεδο δασμολογίου. άρα εδώ πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα μέτρα. μεγάλα σκάνδαλα όπως είδαμε με τη γλυφοσάτη μέτρα αποφασιστικά τα οποία η ευρωπαϊκή ένωση πρέπει να λάβει. ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η πρόταση αυτή δίνει συνέχεια στην πρωτοβουλία των πολιτών κατά της γλυφοσάτης ή στην κατάσταση με το σκάνδαλο της Μοσάντο και τα σχετικά έγγραφα που μας δείχνουν πώς υποβάλλονται μελέτες που ουσιαστικά χρηματοδοτούν οι ίδιες οι επιχειρήσεις ε, θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε τη διαφάνεια και να εξασφαλίσουμε την αντικειμενικότητα και την ανεξαρτησία των επιστημονικών μελετών που χρησιμοποιεί ο Οργανισμός Ασφάλειας Τροφίμων για να χορηγήσει άδειε κυκλοφορία προϊόντων. Θεωρώ ότι το τελικό κείμενο συνιστά σημαντική βελτίωση σε σχέση με την παρούσα νομοθεσία γιατί η αξιολόγηση και η διαχείριση κινδύνων είναι πια μια πιο διαφανής διαδικασία. Ε, Επίση, δημοσιεύονται οι επιστημονικές μελέτες που αποτελούν τη βάση τη αδειοδότηση ε, και μάλιστα δημοσιοποιούνται και οι αιτήσει των παραγωγών. Προβλέπονται και κυρώσεις ε, για παραγωγούς που παραβιάζουν αυτή την ανάγκη της διαφάνειας. Έτσι πιστεύω ότι θα ανακτήσουμε και θα ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Ο αντιπρόεδρο τη Κομισιόν, ο κ. Κατάνιν, έχει το λόγο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την πάρα πολύ καλή συζήτηση και θα ήθελα να επαναλάβω πως η προσωρινή αυτή ε, συμφωνία των συνομοθετών θα ενισχύσει τον σημαντικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο κόσμος θέλει να εμπιστεύεται τις αρχές. και η ΕΦΣΑ πάντα θέλει να εφαρμόζει την ε, αρχή της προφύλαξης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί αν δεν εμπιστευόμαστε τις αρχές... Ε, θα πουλάμε την αλήθεια τελικά. Επίσης, ε, ε, θα ενισχύσουμε την ε, διαφάνεια εδώ πέρα και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω για την καλή δουλειά που κάνετε, για την αποφασιστικότητά σας στο θέμα αυτό και θα ήθελα επίσης ε, να απαντήσω σε κάποια από τα σχόλια για τα προϊόντα που πολλούνται στις αγορές μας. Όλα τα προϊόντα που πολλούνται στις ευρωπαϊκές αγορές πρέπει να ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά κριτήρια ασφάλειας τροφίμων εξαρτήτως προέλευσης. Κάτι το επίσης ε, πολύ σημαντικό. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ασφαλέστερη αγορά και οι προδιαγραφές μας επίσης ισχύουν και για τα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για το ότι σας απασχολούν αυτά τα σημαντικά θέματα. Σας ευχαριστούμε και εμείς κύριε Αντιπρόεδρε. Και τώρα θα ήθελα να δώσω τον λόγο στην εισηγήτρια για δύο λεπτά, την κυρία Πιλάρ Αγιούζο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα απλώς ε, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους ε, που έλαβαν το λόγο, στους και οδησηγητές, να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Κατάινεν και όλους ιδιαίτερως ε, να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες της Επιτροπής και τον Επίτροπο Αντριουκάητες. Παρακαλώ να διαβάσετε τις ευχαριστίες μου και στη Ρουμανική Προεδρία, καθώς και στη συνάδελφο Σόμερ που ξεκίνησε ω πρώτη συγγετήρια αυτή την έκθεση. Και χάρη στη συμβολή όλων αυτών καταφέραμε στη διαπραγμάτευση να καταλήξουμε σε μια σχετικά ικανοποιητική συμφωνία. Οι υπηρεσίες και των τριών οργάνων εργάστηκαν εργοδό τις τελευταίες μήνες και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα κατέληξαν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα. Επίσης, ε, το προσωπικό μας, μας βοήθησε ιδιαίτερω και θα ήθελα και δημοσίω να ευχαριστήσω τους βοηθούς μας. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώνουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. τώρα την επόμενη έκθεση που είναι η έκθεση του κυρίου Λουίς Δεγκράντες Πασκουάλ που αφορά το συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για τα φάρμακα. Θα ακούσουμε πρώτα τον εισηγητή μας, τον κύριο Λουίς Δεγκράντες Πασκουάλ, για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Κατάινεν, για την παρουσία του. Όταν ε, ξεκινήσαμε την εκπάνηση της έκθεσης μου φαινόταν σαν αδύνατη αποστολή. Υπήρχε μεγάλη, ε, μεγάλη διχόνοια στην αρχή, μεγάλος διχασμός και στη ε, διάρκεια των τριμερών ε, διαλόγων καταφέραμε στις 14 ε, Παρθόντος Φεβρουαρίου να καταλήξουμε σε συμφωνία και μάλιστα σε χρόνο ρεκόρ δύο εβδομάδων μετά την αρχική πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θετήθηκε από την πλειοψηφία των κρατών μέλων και επιβεβαιώθηκε και στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και τώρα έφτασε στην Ολομέλεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε αυτό το συμπληρωματικό πιστοποιητικό για να προωθήσει την έρευνα και την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Και η μέση διάρκεια της το διπλώμα του ευρεσιτεχνία είναι τέτοια που δεν αρκεί. Και μάλιστα με αυτό το πιστοποιητικό, το συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασία, επιστρέψαμε τη, ένα τμήμα τη χαμένη προστασία στο διπλώμα του ευρεσιτεχνία. Έτσι όμω αφήσαμε ένα τμήμα τη βιομηχανία ε, ανυπεράσπιστο. Γιατί στη διάρκεια του διπλώματο ευρεσιτεχνία δεν μπορούσε κανεί ε, ούτε να παραγάγει, ούτε να να αποθεματοποιήσει τέτοια προστατευμένα προϊόντα, ούτε καν για την εξαγωγή σε τρίτες χώρες, όσο δεν είχε εκπνεύσει η προστασία. Ενώ για ε, τρίτες χώρες που δεν υπάρχει τέτοια συμπληρωματική περίοδος, υπάρχει δυνατότητα για κάτι τέτοιο. Έτσι, οι παραγωγοί γενοσύμων που θέλουν να εξάγουν εκτός τη Ευρώπη θα έχουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Και μάλιστα ε, τα ευρωπαϊκά γενόσύμα θα προωθούν και στη δική μας αγορά. Είναι σημαντική καινοτομία για τον κλάδο αυτό. Και όταν μιλούμε για τη στρατηγική τη Ευρώπη. θα πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσουμε να υπερασπίζουμε την οικονομία που θα στηρίζεται στη γνώση. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι η βιομηχανία μα αφιερώνει 35 δισεκατομμύρια ευρώ ε, στα θέματα αυτά, στην έρευνα και την ανάπτυξη και εγκρίνονται κάθε χρόνο πολλά νέα φάρμακα και δραστικέ ουσίε. Και μάλιστα ε, τα συστήματα προστασία πνευματική ιδιοκτησία υπάρχουν και λειτουργούν ε, για καινούργια φάρμακα και καινούργιες θεραπευτικές αγωγές. Η βιοφαρμακευτική βιομηχανία των ε, γενώσιμων προϊόντων θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις αξιαγωγές μας και να αποτελέσει ακοργωνιαίο ολίθο της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, ώστε να ανακάψουμε πολύ πιο γρήγορα. Η παράταση του πιστοποιητικού εξασφαλίζει μια ε, ισοτιμία στο πλαίσιο αυτό μεταξύ των παραγωγών γενοσύμων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των παραγωγών γενοσύμων τρίτων χωρών. Αυτή, από τώρα η παραγωγή γενοσύμων και βιομοειδών που ε, έχουν έμπρεπε την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούν να εξάγουν προϊόντα αυτά σε χώρες που έχει εκπνεύσει το πιστοποιητικό και ακόμη και αν καλύπτονται από συμπληρωματικό ε, πιστοποιητικό προστασία στην αγορά. Επίση, οι ίδιοι παραγωγοί θα μπορούν να αποθεματοποιούν τα προϊόντα στη χώρα που παρήγαν, τα, κατά το τελευταίο εξάμεινο της, της ισχύω προστασίας και μετά την εκπνοή του πιστοποιητικού θα βοηθήσουμε τη βιομηχανία να είναι πιο ανταγωνιστική ε, αμέσως μετά την εκπνοή του πιστοποιητικού. Επίσης, έχουμε και ασφαλιστικές δεκλίδες για να μην παραβιάσουμε την πνευματική ιδιοκτησία την καινοτομία. Και γι' αυτό απαιτούμε από, την από τους παραγωγούς και βιομοιδών προϊόντων να δημοσιοποιούν και να ενημερώνουν τον κάτοχο του συμπληρωματικού πιστοποιητικού και μάλιστα με τρεις μήνες προθεσμία. Με την, ειδοποίηση αυτή, με την κοινοποίηση αυτή θα έχουμε διαφανές συστήμα και θα εξασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών αγορών. Ταυτόχρονα ο κανονισμός ε, κρατάει εμπιστευτικέ τις πιο ευαίσθητες πληροφορίες. Η έγκριση του κανονισμού αυτού θα ευνοήσει ιδιαίτερως ε, την ε, ευρωπαϊκή βιομηχανία και μάλιστα το 2025 θα έχουμε αύξηση της παραγωγής από 7,5 με 9,5 δις και θα δημιουργηθούν περίπου 20 με 25.000 θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έχουμε εξοικονομήσεις στις φαρμακευτικές δαπάνες περίπου 4%. Δεν ήταν εύκολη έκθεση. Όλοι χρειάστηκε να κάνουμε προσπάθειες και παραχωρήσεις για να καταλήξουμε σε συμφωνία και ισορροπία. Και ευχαριστώ και τους και ηγητές. Ευχαριστώ τους συνεργάτες μας που ε, εργάστηκαν άοκνα, κυρίως τη δική μου βοηθό, τη Μερσέδες, που εργάστηκε εργοδός και ευχαριστώ και την Ρουμανική Προεδρία που έδωσε προτεραιότητα σε αυτό το σημαντικό θέμα. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Εξ ονόματος της Κομισιόν. Κύριε Κατάινεν, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ. η απαλλαγή από συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασία ήταν σημαντικό κομμάτι τη κοινή αγορά και σημαντικό παραδοτέο στόχο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήταν κάτι το οποίο είχε ζητηθεί ρητά στην έκθεση τη κυρία Λάρα Κόμι του 2016 για τη στρατηγική τη κοινή αγορά. Μια θετική ψηφοφορία αύριο θα στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στου Ευρωπαίου πολίτε και στι επιχειρήσει. Ένα θετικό μήνυμα για την ανταγωνιστικότητα ένα θετικό μήνυμα για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και για την πρόσβαση σε φτηνά φάρμακα. Το να έχουμε λοιπόν αποτελέσματα για τους πολίτες μας ε, είναι κάτι σημαντικό, όπως και το να φαίνεται άλλωστε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό λοιπόν να το καταφέρουμε μέχρι τον επόμενο μήνα. Η Κομισιόν είναι πολύ ικανοποιημένη από, από την έκβαση των διαπραγματεύσεων το Κοινοβούλιο και η Ρουμανική Προεδρία έκαναν εξαιρετική δουλειά, κυρία Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ. Δεν ήταν εύκολη η δουλειά στο θέμα αυτό. Κάθε άλλο. Οπότε θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Ντεγκάντε Πασκουάλ, για την ε, άοκνη εργασία του. Υπό δύσκολε συνθήκες. Θα ήθελα επίση να ευχαριστήσω τους κυρίους Βίλκεν και Σάντσες και τους λοιπούς ε, σκιώδεις εισηγητές. Ε, με την δουλειά που κάνατε συνεισφέρατε σε μια οικονομικά χρήσιμη ε, απαλλαγή και σε ένα ισορροπημένο και σαφές νομικό κείμενο. Το κείμενο αυτό το οποίο συμφωνήσατε με το Συμφούλιο θα επιτρέψει σε ευρωπαϊκές εταιρείες να γίνουν ηγέτες στην παγκόσμια αγορά των γεννόσιμων φαρμάκων και να κινούνται με ίσους όρους με τις εταιρείες που έχουν την έδρα τους ε, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναμένουμε τη δημιουργία 25.000 θέσεων εργασίας τα επόμενα χρόνια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως το να εδρεωθεί η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως κόμβος Έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας. Θα αναφέρω τώρα ορισμένα πράγματα ε, για τον κανονισμό που θα ψηφιστεί αύριο. Πρώτα απ' όλα για τα αποθέματα, ένα ευαίσθητο ζήτημα για το Κοινοβούλιο. Καλωσορίζω την ευελιξία που επέδειξε το Συμβούλιο και η Κομισιόν στο να δεχτεί τη συμπερίληψη αυτή. Θα επιτρέπεται η δημιουργία αποθεμάτων κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών ε, για να διασφαλιστεί καλύτερα η ομαλή μετάβαση μετά την πρώτη μέρα ε, μετάβαση των νέο καθώς μετά την λήξη δηλαδή του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας και κατόπιν μετά από ε, κάποια χρόνια η Κομισιόν θα λάβει υπόψη το εάν είναι ικανοποιητικέ συνθήκε στην αγορά. Πλέον, η ρήτρα αναθεώρηση στο αρθρο 21 21α του κανονισμού λέει πω η Κομισιόν θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη μεταξύ άλλων το εάν η περίοδο ε, αποθεμάτων έξι μηνών επαρκεί για να εκπληρωθούν οι στόχοι. Δεύτερον, και τα τρία θεσμικά όργανα επέδειξαν ευελιξία. Οπότε η κατάρριξη του του πιστοποιητικού προστασία θα γίνει πραγματικότητα το 2022 το αργότερο. Έτσι λοιπόν σεβόμαστε τους δύο, δύο στόχους. Το να είναι και νομικά σωστή και οικονομικά χρήσιμη. Τούτου λεχθέντος δεν θα υπάρχει ε, αναδρομικότητα. Παρομοίως τα δικαιώματα των κατόχων συμπληρωματικών πιστοποιητικών προστασίας δεν επηρεάζονται καθώ παραμένουν ε, τα ίδια κατά τη διάρκεια ισχύω των πιστοποιητικών. Επιπλέον θα υπάρξει ένα μεταβατικό καθεστώς το οποίο λαμβάνει υπόψη τις θεμητές προσδοκίες των κατόχων των δικαιωμάτων. Τρίτον, για τις δικλείδες ασφαλεία, ε, Ο τελικός συμβασμός είναι εύρωστος και με διαφάνεια εξαιρέσεις ε, θα έχουν ε, σημαντικές ε, και αναλογικές δικλείδες ασφαλείας μεταξύ των οποίων η ειδοποίηση που σχετίζεται και με τους κανόνες που θα τεθούν ενισχύ, που τα ετέθησαν ενισχύ τον Φεβρουάριο του 2019. Ταυτόχρονα όμως ο σεβασμός σέβεται τις ανάγκες των κατασκευαστών γενοσύμων φαρμάκων για να μπορέσουν να διατηρήσουν την εμπορική τους για να μπορέσει να συνεχίσει η πορεία του και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παραπέρα, γιατί αυτό μακροπρόθεσμα σημαίνει χαμηλέ τιμέ για του ασθενεί. Τέλο, θεωρώ ότι επιτύχατε έναν καλό συμβιβασμό. Αποτελεί μια καλή ισορροπία μεταξύ των διάφορων πολιτικών απόψεων και των ε, διαφορετικών συμφερόντων και ελπίζω το Κοινοβούλιο να την εγκρίνει στην αυριανή ψηφοφορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Βέλκεν για την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια, τον εισηγητή για την πολύ καλή συνεργασία και τους υπόλοιπους συναδέλφους γιατί πρόκειται για κάτι το πολύ δύσκολο. Τι πετύχαμε τώρα εδώ με αυτή την έκθεση. Θεωρώ ότι διασφαλίζουμε το ότι οι ασθενείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουν καλύτερη πρόσβαση σε φτηνότερα και ασφαλή φάρμακα. Θεωρώ ότι με αυτόν τον ε, τρόπο καταφέραμε επιτέλους να εκπληρώσουμε την εντολή που είχε δοθεί σε διάφορες εκθέσεις του Κοινοβουλίου. Δηλαδή θα έχουμε στην Ευρώπη γενώσιμα βιομοειδή ε, φάρμακα. Έτσι αυξάνεται η ασφάλεια για τους ασθενείς ε, και θυμόμαστε ότι τα τελευταία χρόνια υπήρχαν κάποια φάρμακα τα οποία δεν ήταν σωστά παρασκευασμένα, υπήρχε σπάνις άλλων ε, φαρμάκων, έτσι μπορούμε να φροντίσουμε ότι θα υπάρχουν επαρκή αποθέματα. Ποιο είναι λοιπόν το επίμαχο σημείο εδώ πέρα ήταν τα αποθέματα για τις πρώτες ημέρες μετά την λήξη του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας. Και εδώ πέρα, σε μεγάλο βαθμό εντός του Κοινοβουλίου, αλλά δυστυχώς και η Κομισιόν, καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια για να μην υπάρξει απόθεμα και αποθεματοποίηση. Και παρά το ότι η μελέτη αντικτύπου της ίδιας Κομισιόν λέει ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για κάτι τέτοιο. Υπάρχει συγκεκριμένα στην, στο σημείο 42 της ε, μελέτης αντικτύπου. Τελικά είχαμε ένα απόθεμα έξι μηνών που καταφέραμε να περάσουμε και μέσω της ρήτρα αναθεώρησης έχουμε την δυνατότητα να δούμε κοντά στα γεγονότα εάν πραγματικά επαρκεί κάτι τέτοιο για να έχουν επαρκή φάρμακα όλοι οι ασθενείς. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω και εσάς και όλους τους συνεργάτες που εργάστηκαν μεγάλη πίεση χρόνου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Λοτόφσκι κατόπιν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή. Ο συγκεκριμένος κανονισμός ε, είναι από τα λίγα παράδειγματα που το ευρωπαϊκό δίκαιο μπορεί να είναι θετικό, ακόμη και για την Πολωνία. Και σπάνια είχαμε στην παρούσα κοινοβουλευτική θητεία τόσο ευνοϊκές νομοθετικές προτάσεις. Και φυσικά θα ε, βοηθήσουμε τους παρασκευαστές προϊόντων και θα βοηθήσουμε και τους ασθενείς. Είναι πολύ καλό το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ανοίγουν νέες αγορές και μεγάλες προοπτικές για τους Ευρωπαίους παρασκευαστές ε, γενώσιμων και βιόμοιδων ε, προϊόντων. Είναι επίσης θετική νομοθεσία και για τους ε, ασθενείς που θα έχουν πρόσβαση σε καινοτόμα και αποτελεσματικά φάρμακα. νομίζω ότι η βιομηχανία θα αξιοποιήσει την ευκαιρία του κανονισμού ε, θα δημιουργήσει νέες θέσει απασχόλησης σε αυτό το καινοτόμο τομέα της βιομηχανία και φυσικά η ομάδα μου θα υποστηρίξει αύριο τη σχετική έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βίρινγκ για 1,5 λεπτό έχει το λόγο εκ μέρου τη Άλτα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στην ομιλία αυτή θα τονίσω πως υπάρχει το επίκεντρο είναι ο ασθενής και η φαρμακοβιομηχανία. Για εμένα αυτό το οποίο έχει πρώτη σημασία είναι τα συμφέροντα των ασθενών και έχω βεβαίως ήδη απειρά γιατί έχω επιζήσει από τον καρκίνο. Θα πρέπει λοιπόν η Κομισιό να ξαναδεί τα πράγματα και να παραμείνει εντός ορίων. Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ε, των ε, φαρμακευτικών εταιριών είναι άμοιβη για την έρευνα που κάνουν επί σειρά ετών για να μπορέσουν τελικά να βγάλουν ένα φάρμακο στην αγορά. Μίλησα βεβαίως για άμοιβη, θα έπρεπε μάλλον να το πούμε ασφάλεια. Οι επιχειρήσεις οι οποίες ε, Ε, επενδύουν στην έρευνα ξοδεύουν τεράστια ποσά. Παραδείγματο χάρη για ένα νέο αντιβιωτικό. Θα είναι επιτυχημένο μόνο ένα στα 10.000 μόρια τα οποία δοκιμάζονται. Βεβαίω θα πρέπει ε, και από αυτά να αναπτυχθούν αρκετά σε έναν αρκετά μεγάλο βαθμό για να καταλήξουν να δουν ποιο τελικά λειτουργεί. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τα δικαιώματα ευρεστιχνίας και με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησία. Δεν θα πρέπει λοιπόν να ξεχνάμε τις πιθανές συνέπειες που μπορεί να πλήξουν τον κλάδο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Τον λόγο έχει τώρα η κυρία Κονέτσνα για την ΚΟΕ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, τη στιγμή αυτή οι παρασκευαστές γενώσιμων και βιομοειδών ε, φαρμάκων που έχουν έντρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν να παρασκευάσουν φάρμακα και να τα εξάγουν στις τρίτες χώρες ακόμη και σε περίπτωση που έχει εκπνεύσει η προστασία του προϊόντος. Και έτσι χάνουμε πολλές θέσεις απασχόλησης, αλλά και προς, ε, μειώνεται η πρόσβαση σε καινοτόμα και αποτελεσματικά φάρμακα. Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος προσπαθήσαμε να βρούμε μια ισορροπία ε, στο κείμενο αυτό. Ε, και το αποτέλεσμα δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό. Το πρόβλημα που διαπιστώνω εγώ στην έκθεση αυτή είναι η θέση σε ισχύ του κανονισμού και από πότε μπορούν ε, οι ασθενείς να υποφεληθούν από το κανονισμό. Νομίζω ότι είναι υπερβολική η μεταβατική προθεσμία των τριών ετών. Έπρεπε αμέσως οι ασθενεί να μπορούν να αποφελούνται από τις νέες διατάξει Επίσης θα πρέπει να προστατεύσουμε περισσότερο στο μέλλον τους παρασκευαστές ε, γενώσιμων και ομοειδών, ε, βιομοειδών φαρμάκων. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρέντα, εκ μέρους των Πρασίνων. Σήμερα είναι η τελευταία μου ομιλία σε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είμαι υπερήφανη που η ομιλία μου γίνεται σε ένα χαρτοφυλάκι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κινήθηκε ε, στα, κατά εκείνων της βιομηχανίας των πνευματικών δικαιωμάτων που βάζουν τα κέρδη πάνω από την ασφαλή πρόσβαση στα φάρμακα. Δεν είναι οικονομικά, αυτά τα πιστοποιητικά παρατείνουν τα πνευματικά δικαιώματα σε φάρμακα που ήδη έχουν μακροχρόνια άδεια. Αυτή η πρόταση επιτρέπει τουλάχιστον να παρασκευάζονται γενώσιμα για πωλήσει όπου εκεί ήδη είναι νόμιμα. Αυτό είναι ένα μικρό βήμα, αλλά είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και έρχεται με φιλόδοξη ρήτρα αναθεώρηση για να εξηχνιαστεί κατά πόσο αυτή η εξαίρεση για έξι μήνε για την αποθήκευση αρκεί για να επιτευχθούν οι στόχοι δημόσια υγεία. Είναι χρειαζόμαστε να αμφισβητήσουμε το καθεστώ για αυτέ τι άδειε, τι συμπληρωματικέ και να έχουμε πιο θεμελιώδη μεταρρύθμιση. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και τα ξαναλέμε στο Ιπανιδί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Μπουσόλ, Πέτερλε, ο κ. Σαλό και ο κ. Μαριά. Πρώτα είναι ο κ. Μπουσόη που θα πάρει το λόγο. Στα πλαίσια τη διαδικασία Catch the Eye. Ευχαριστώ. Πολύ σημαντικό ο κανονισμό που δίνει εξαίρεση στι ε, ε, βιομηχανικές, ε, ευρωπαϊκέ βιομηχανίε που μπορούν να παρασκευάσουν αβιανόσημα και βιομοειδή μόνο για εξαγωγή προ τρίτε χώρε ε, για τις οποίες έχει λήξει το πιστοποιητικό προστασίας και μπορούν να τις αποθεματοποιούν, αποθεματοποιούν τα, τα φάρμακα αυτά από την πρώτη μέρα εκπνοής ε, του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας. Έτσι, οι παραγωγοί μας θα γίνουν ανταγωνιστικοί στις αγορές τρίτων χωρών όπου η συμπληρωματική προστασία είτε δεν υπήρχε είτε έχει εκπνεύσει, αλλά και εξασφαλίζει πρόσβαση εγκαίρως στους πολίτες μας ε, σε φάρμακα μειωμένης τιμής ενώ γνωρίζουμε πόσο υψηλέ είναι οι τιμέ των φαρμάκων και μερικέ φορέ δυσβάσταχτε για του ασθενεί. Ευχαριστώ τον εισηγητή, τον κύριο Στεγκράντε Πασκουάλ, για την εξαιρετική του προσπάθεια και την πολύ έκθεση. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Ο κύριο Μαριά τώρα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι το βασικό θέμα που συζητούμε και στο οποίο πρέπει να επικεντρωθούμε είναι η προστασία της δημόσιας υγείας δεύτερον το συμφέρον των ίδιων των ασθενών που αυτό προϋποθέτει πρόσβαση των ασθενών σε φθηνά φάρμακα. επομένως οι όποιες ρυθμίσεις γίνονται για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής φαρμακοβιομηχανίας πρέπει να υπηρετούν αυτούς τους στόχους διότι δεν πρέπει να φτάσουμε στο άλλο άκρο να έχουμε δηλαδή ακριβά φάρμακα στα οποία να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση οι ασθενείς διότι ξέρουμε ότι έχουν γίνει διάφορα τρίκ από τις φαρμακευτικές στην ευρώπη προκειμένου να ανεβάσουν την τιμή του φαρμάκου. κλασική περίπτωση το σκάνδαλο Novartis, το οποίο έχει αποκαλυφθεί ιδίως στην ελλάδα και για το οποίο πρέπει να πάμε μέχρι το τέλος να αποκαλυφθούν όλες οι ευθύνες και φυσικά να επιβληθούν ποινές και στη συγκεκριμένη φαρμακοβιομηχανία πρέπει να προσέξετε κύριε επίτροπε κυρία κατάινεν το θέμα των αποθεμάτων σε φάρμακα διότι αυτό είναι βασικό όπως επίσης να μην αξιοποιούν οι πολυεθνικές την ευκαιρία για εξαγωγή των φαρμάκων και να έχουμε έλλειψη μέσα στην ευρωπαϊκή ένωση. αν τηρήσουμε όλα αυτά τότε μπορούμε να έχουμε και ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής φαρμακοβιομηχανίας αλλά κυρίως προστασία των ασθενών. ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. köszönjük, és Alois következik. Parancsoljon Ευχαριστώ. Ο Αλόης Πέτερλε έχει τώρα τον λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Κύριε Αντιπρόεδρε της ε, Κομισιόν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ντεγκράντες Πασκουάλ για τη δουλειά που έκανε Ανοδεχούμενη η αλλαγή της ε, νομοθεσίας όσον αφορά το συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας. Ε, κερδίσαμε πολλά εδώ πέρα. Θα έχουμε καινούργια φάρμακα στην Ευρώπη και ίσως όρους ανταγωνισμού για τους ε, παραγωγούς γενοσύμων και βιομοιδών στην Ευρώπη. Ε, των εταιριών δηλαδή που έχουν έδρα στην Ευρώπη σε σχέση με αυτούς που έχουν έδρα σε τρίτες χώρες και έτσι θα κάνουμε και εξαγωγές και επίσης ε, το κάναμε και πιο εύκολο να υπάρχει είσοδο στην ευρωπαϊκή αγορά την επομένη της λήξης του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας. Τα τελευταία χρόνια το κόστος ε, έχει αυξηθεί πάρα πολύ Πρέπει να φροντίσουμε να φτάνουν τα φάρμακα στην αγορά γρηγορότερα και αυτό σημαίνει ότι οι ασθενείς θα έχουν γρηγορότερη πρόσβαση σε φτηνότερα φάρμακα. Άλλη μια απόδειξη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται για τους ασθενείς και λειτουργεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να ολοκληρωθεί η συζήτηση θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον Αντιπρόεδρο της Κομισιόν, κύριο Κατάινεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Θέλω να ευχαριστήσω για την καλή αυτή συζήτηση. Ευχαριστώ εκ νέου και συγχαίρω τον εισηγητή. Πολύ καλή δουλειά έκανε. Υπήρξε πολιτικά ευαίσθητο θέμα, αλλά δείχνει ρεαλισμό η λύση. Πολύ πρακτική λύση που εξευρέθη. Δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πληρ... εξασφαλίζει ότι είναι στα ίδια επίπεδα η παραγωγή βιομοειδών ή ε, γενοσύμων όπως και άλλοι. Ταυτόχρονα, η προστασία του διπλώματος ευστεχνίας ε, και των πνευματικών δικαιωμάτων καλύπτει εκείνους που ανακαλύπτουν καινοτομίε. Αυτή είναι η περιγραφή της συμβαστικής λύσης. Αυτά πετυχαίνει. Θα δείξουμε έτσι σε αυτούς που καινοτομούν ότι αυτή η Ήπειρος υποστηρίζει την καινοτομία, ότι θέλουμε να προστατεύσουμε και ότι ταυτόχρονα δημιουργήσαμε ισότιμους όρους για εκείνους που παράγουν τα γενώσιμα και τα βιοομοειδή. Πολύ καλή απόφαση, λοιπόν, για τους ασθενείς μας, για τους καταναλωτές και πολύ καλή απόφαση και για τη βιομηχανία και τους καινοτόμους, αυτούς που παράγουν τα φάρμακα. Ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία σας. Ευχαριστώ πολύ για αυτά που είπατε, κύριε Επίτροπε. Και τώρα να δώσω το λόγο στον εισηγητή μα για να ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση. Δύο λεπτά έχετε στη διάθεσή σα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρουσία σας, για τα λόγια σας, ε, για το σθένο σας και ευχαριστώ και τους κοιόδης ηγετές. Μερικές φορές στη διαδικασία των συζητήσεων ένιωσα μοναξιά, γιατί οι σκιώδεις ηγητές παρά ήταν απαιτητικοί απέναντί μου, αλλά καλά έκαναν απέτησαν την επίτευξη ισορροπίας και συμβαστικής λύσης. Μερικές φορές αναζητώντας συμβιβασμό έχουμε μια σχετικά κακή λύση, κακό αποτέλεσμα. Ότι είναι όρο και έτσι και εμεί μερικέ φορέ. Αλλά, μην, δεν, θα, δεν είναι η συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί παρά του συμβασμού καταλήξαμε σε ισορροπημένο αποτέλεσμα. Και έτσι και προσπίζουμε τα θεμήτα συμφέροντα των ε, παρασκευαστών ε, γενώσιμων και βιομοειδών φαρμάκων, αλλά ταυτόχρονα προστατεύουμε και την δημόσια υγεία και τα δικαιώματα του ασθενούς. Και ακριβώς επειδή κρίναμε ότι μπορεί στο μέλλον να αποδειχθεί ότι δεν είναι αρκετό ο κανονισμός, προβλέψαμε και αυτή τη ρήτρα αναθεώρησης. Νομίζω ότι εκπληρώσαμε του στόχου μα ε, σε αυτή την κοινοβουλευτική θητεία, από την οποία και εγώ αποχωρώ και δεν πρόκειται να ξαναγυρίσω και ευχαριστώ για τη συνεργασία που είχαμε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πασκουάλ, ευχαριστώ για τη συζήτηση. Πέρα η συζήτηση, η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο. Ευχαριστώ πολύ για το έργο σας και καλωσορίζω την, καλή, την κυρία Γιούροβα. Κύριε Κατάιναν, ευχαριστώ πολύ. Και τώρα φτάνουμε στο επόμενο σημείο, στο επόμενο θέμα μας, δήλωση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενδεχόμενη έκδοση του Τζούλιαν Assange. Καλωσορίζω ε, Λοιπόν, την κυρία Σιώτα, έχετε το λόγο. Αξιότιμα μέλη, επίτροπε κυρία Γιούροβα, ευχαριστώ για την ευκαιρία να συζητήσουμε το θέμα της ενδεχόμενης έκδοσης του Τζούλιαν Ασάνς. Όλοι γνωρίζουμε ότι όταν ενεργεί κανείς για προστασία των ε, δημοσίων συμφερόντων, οι καταγγέλλοντες παίζουν σημαντικό ρόλο για να καταγγέλουν διάφορες ε, παράνομες ενέργειες και γι' αυτό ε, χρήζουν παράνο... προστασίας νομικής. Το συζητήσαμε αυτό χθες στην συζήτηση που είχαμε για την οδηγία για τους καταγγέλλοντες. Όλοι παρακολουθούσαμε τα πρόσφατα γεγονότα που σχετιζόταν με τον κύριο Ασάνς. Ο Τζούλιαν Ασάνς κατέφυγε στην πρεσβεία του Εκουαδόρ στο Λονδίνο το 2012 για να αποφύγει να απελαθεί στην Σουηδία για να δικαστεί για βιασμό και διάφορα, διάφορες άλλες κατηγορίες. Έλεγε ότι το ήθελε να αποφύγει να εκδοθεί στη ΣΥΠΑ και να δικαστεί γιατί δημοσίευσε χιλιάδε επί χιλιάδων ε, πλαστογραφημένα έγγραφα των ΗΠΑ. Στις 11 Απριλίου το Εκουαδόρ απέσυρε το άσυλο του κυρίου Ασάν και αυτό οδήγησε στη σύλληψή του από τη Βρετανική αστυνομία. Το δικαστήριο του Westminster ακολούθω, τον βρήκε ένοχο για κατηγορίες των Βρετανών για παραβίαση της εγγύσης με την οποία έχει απελευθερωθεί. Πέρα από τι κατηγορίε του Ηνωμένου Βασίλειου, ο κ. αντιμετωπίζει και κατηγορίε και στι Ηνωμένε και οι Σουηδικέ δικαστικέ αρχέ ανέφεραν ότι οι έρευνε που αφορούν το άτομό του ίσω οδηγήσουν να απαγγελθούν εκ νέου κατηγορίε για βιασμό. Να πω ότι το Συμβούλιο αυτό κάθε αυτό δεν έχει συζητήσει το ζήτημα του κυρίου Ασάνς και το ενδεχόμενο έκδοσή του και δεν έχει κάποια θέση από αυτού. Είναι γεγονός ότι οι εκδόσεις είναι θέμα αποκλειστικής αρμοδιότητας ε, των κρατών μελών. Γι' αυτό το θέμα τώρα βρίσκεται στα χέρια του Βρετανικού δικαστικού κλάδου και ε, του Υπουργού Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου. Δράτω με τη ευκαιρία όμω να τονίσω εκ νέου ότι το Συμβούλιο προσδίδει πολύ μεγάλη σημασία στην προστασία των κατακέλλοντων είναι γεγονός κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εστιάστηκαν επί του, της εξασφαλίσεως συμφωνίας όσον αφορά την οδηγία για τους καταγγέλλοντες και να καταλήξουμε συμφωνία πριν ε, ολοκληρωθεί αυτή η θητεία. Αυτός ο στόχος επετεύχθη και αυτή η Ολομέλεια ψήφισε σήμερα το κείμενο που συμφώνησαν οι διαπραγματευτές των δύο συνομοθετικών κλάδων. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ για αυτά που μας είπατε, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον λόγο τώρα έχει η κυρία Γιούροβα εξ ονόματος της Κομισιόν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μας ζήτησε να κάνουμε μία δήλωση για την πιθανή έκδοση του Τζούλιαν Νασάντζα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Μπορούμε να σας ενημερώσουμε πως η έκδοση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών ε, βασίζεται σε διμερή συνθήκη και Συμφωνία Έκδοσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν επιτρέπεται η έκδοση στην περίπτωση που υπάρχουν λόγοι να υποψιαζόμαστε, να θεωρούμε ότι μπορεί να υπάρξει εφαρμογή της ανατικής ποινής. Επιπλέον λέγεται πως το κράτος μέλος δεν θα πρέπει να προχωρήσει έκδοση εάν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων του υπόπτου στην περίπτωση που η Σουηδία αποφασίσει να εκδώσει νέο ευρωπαϊκό ένταλμα μετά από αυτό το οποίο είχε ανακαλέσει το 2017 και το Βρετανικό Δικαστήριο θα έπρεπε να εξετάσει το εάν θα προηγηθεί το ε, ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης ή το αμερικανικό ένταλμα έκδοσης. Δεν υπάρχουν σαφείς κανόνες, αλλά κάποιοι παράγοντες που θα λάβει υπόψη το δικαστήριο. Ως γενική παρατήρηση πρέπει να σημειώσω πως η Κομισιόν δεν έχει αρμοδιότητα για να παρέμβει σε δικαστικές διαδικασίες που εκκρεμούν στα δικαστήρια των κρατών μελών. Βασιζόμαστε πλήρως στην ανεξαρτησία και τον επαγγελματισμό των Βρετανικών δικαστηρίων για να λάβουν την σωστή απόφαση, ε, καθώς έχουν και μπροστά τους τα στοιχεία. Σας ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο πρώτος ομιλητής είναι ο κύριος Πόσπισιλ για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να συμφωνήσω με την Επίτροπο και να πω και εγώ ότι δεν καταλαβαίνω γιατί συζητούμε την υπόθεση αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε μια συγκεκριμένη υπόθεση αιτήματο έκδοσης που θα εκδικαστεί με βάση τις διεθνείς συμφωνίες. Έχουμε την δικαιοδοσία του Ηνωμένου Βασιλείου, έχουμε τις Ηνωμένε Πολιτείε που ζητούν την έκδοση. Πρόκειται για δύο κράτη δικαίου και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η δικαστική διαδικασία θα είναι απόλυτα σωστή με τις κατάλληλες οικονομικές ε, εγγυήσεις και με σεβασμό του κράτους δικαίου. Μπορούμε να συμφωνούμε ή να διαφωνούμε με τις ενέργειες του κυρίου Ασάνζ. Εγώ διαφωνώ. Θεωρώ ότι η ελευθερία έκφρασης έχει τα όρια του και δεν μπορεί να, και να παραβιάζει το ε, απόρριτο, το εθνικό ή τους όρους εθνικής ασφάλειας. Αλλά Σίγουρα οι αρμόδιες δικαιοδοσίες θα πρέπει να αποφασίσουν για την υπόθεση Ασάνς και είναι σωστό που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι οι πολιτικές αρχές δεν δικαιούνται να επεμβαίνουν στο δικαστικό σύστημα, στη δικαστική εξουσία μιας άλλης χώρας. Ας αφήσουμε το ζήτημα στα Βρετανικά δικαστήρια, στους Βρετανούς δικαστές που θα εκδικάσουν το αίτημα της έκδοσης και θα κρίνουν αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την έκδοση του κυρίου Ασάνς στις Ηνωμένε Πολιτείε. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο Βρετανικό δικαστικό σύστημα. Ευχαριστώ κυρία Γκόμες εκ μέρους Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Η έκδοση του Ζουλίαν σας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ε, θα πρέπει να παρεμποδιστεί. Μόνο έτσι θα εξασφαλίσουμε ε, προστασία της Ευρώπης όποιον θέλει διαφάνεια και, προσ... και ε, προασπίζει την αλήθεια όταν μια κυβέρνηση σαν το Τραμπ που, που χρησιμοποιεί τα ΜΜΕ για τους δικούς στόχους δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε την έκδοση του Ασάνς γιατί ο κύριος Τραμπ ε, εργαλειο, έχει εργαλειοποιήσει αυτό το θέμα και ο Ασάνς θα διέτρεχε κίνδυνο να καταδικαστεί ακόμη και στην ασχάτη των ποινών όπως ε, επισημαίνουν σημαντικές οργανώσεις ε, ε, πίεσης, προστασίας δικαιωμάτων. Είδαμε τι έγινε με την περίπτωση του Μάνικ που υπέστη και βασανιστήρια ε, για την ε, καταγγελία κάποιων στοιχείων. Είδαμε τι έγινε στο Γουαντάναμο και στις μυστικές φυλακές. Είναι τρομερή η υποκρισία των Αμερικανών και των συνένοχων μερικές φορές ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Ε, και μάλιστα ένας υπουργό που με καταδίκασε ε, όταν ζήτησα διερευνητική ε, επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να εξετάσουμε τις μυστικές πτήσεις στην Πορτογαλία και σε μυστικές φυλακές από το Γουαντάναμο. με κατηγόρησαν ότι προσπίζω τον ιδρυτή του Wikileaks. Θα πρέπει λοιπόν αν όντως διέπραξε κάποια αδικήματα ο κύριος Ασάνζ να δώσει λόγο στα σουηδικά δικαστήρια που δίνουν τις δικονομικές εγγύσεις για τη δίκαιη δίκη αλλά να μην γίνει η έκδοσή του προς τις Ηνωμένε Πολιτείες. Με ανησυχεί ιδιαίτερος που ε, ο Ζούλιαν Ασάνζ παραδόθηκε από την ε, πρεσβεία του Ισημερινού από μια χώρα που συνεργάστηκε με τον Πούτιν για να επέμβει στις αμερικανικές εκλογές. Και είδαμε τι έγινε με την ειδική περίπτωση του Μίλλερ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα πρέπει λοιπόν να εγγυηθούμε δικαιοσύνη και δίκαιη δίκη στον Ζουλιαν Ασάνζ. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τον Ασάνζ, να προστατεύσουμε τους ε, καταγγέλλοντες και να εγγυηθούμε τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες. Ε, να προστατεύσουμε αυτούς που διακινδυνεύουν τη ζωή τους για την ελευθερία και τη διαφάνεια. Ο Ζουλία Σάνζ αξίζει την προστασία μας και αξίζει να απολαύσει όλα αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δέχεστε μια γαλάζια κάρτα από τον κύριο Πόσπισιλ. Κύριε Πόσπη, συλλέχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφε, παρακολούθησα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ε, την παρέμβασή σα. Είμαι πρώην Υπουργό τη Δικαιοσύνη και σα ερωτώ το εξή. Πώ είναι δυνατό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομοθετική εξουσία να επεμβαίνει σε μία δικαστική υπόθεση. Μιλούμε για μία διαδικασία έκδοσης ε, ε, είναι μια υπόθεση που απασχολεί τα δικαστήρια. Εμεί είμαστε πολιτικοί. Δεν μπορούμε να προστατεύουμε εμεί ω πολιτικοί ε, κάποιον όπω ε, προτείνατε, κάποιον που ενέχεται σε μια διαδικασία έκδοσης. Πώς το δικαιολογείτε. Κοιτάξτε, δεν πρέπει καμία ευρωπαϊκή χώρα να κάνει εκδόσει προ μια χώρα που έχει τη θανατική ποινή και αυτό ισχύει για τι Ηνωμένες και λυπάμαι γι' αυτό. Και πράγματι ο Ασάντ, αν εκδοθεί στι Ηνωμένε Πολιτείε, μπορεί να μετωπίσει κατηγορία για κατασκοπία που συνεπάγεται θανατική ποινή. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ε, νομικό και πολιτικό λόγο για τον οποίο δεν πρέπει να εκδοθεί από ένα δικαστήριο είτε στον Ηνωμένο Βασίλειο, είτε στη Σουηδία, είτε στη δική σα χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενο, ο κ. Ουρμπαν Κρέσπο, εκ μέρου τη ΓΚΟΕ. Ευχαριστώ. Η κράτηση του Ασάνς σηματοδοτεί μια πολύ σκοτεινή στιγμή για την ελευθερία της έκφρασης. Η σύλληψη και κράτησή του μας ε, αγγίζει όλους και τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν χάρη στον Ασάνς και το Wikileaks ε, αποκάλυψαν δολοφονίες δημοσιογράφων, ε, πολλοί άριθμες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο και η ομάδα εργασίας για τις αυθαίρετες κρατήσεις έκρινε παράνομη την κράτηση του Ζούλια Ρασάνς. Επίσης, έχουμε κρούσει το κόδωρο του κινδύνου για την έκδοση του ΑΣΑΝ στι ε, Ηνωμένε Πολιτείε. Σήμερα εγκρίναμε οδηγία για την προστασία των πληροφοριοδοτών. Θα πρέπει να την τηρήσουμε. Η έκδοση του ΑΣΑΝ θα έδινε ένα πολύ επικίνδυνο μήνυμα. Θα έδινε το μήνυμα ότι αυτοί που ψώνουν το παράστημά τους ε, απέναντι στη διαφθορά, στην κατάχρηση εξουσίας, το πληρώνουν με το κεφάλι του. Αν τον εκδώσουμε στι Ηνωμένε Πολιτείε, ουσιαστικά θα απαρνηθούμε θεμελιώδε τμήμα τη δημοκρατία μα. Θα απαρνηθούμε το αναπαλωτρίο, το δικαίωμα στην ελευθερία έκφραση. Α μην το επιτρέψουμε, κυρίε και κύριοι. Σα ευχαριστώ. Τον λόγο έχει η κυρία Εύα Ζολή. Η ενδεχόμενη έκδοση του Ζούλιαν Ασάν, του ιδρυτού του Wikileaks, προ τι Ηνωμένε Πολιτείε, είναι κάτι που δεν αφορά τη μοίρα ενός ανθρώπου, αλλά αγραφούμε έτσι και το μέλλον των δημοκρατιών μας. Θα πρέπει να επερασπιστούμε με κάθε προσπάθεια την ελευθερία τη ενημέρωση, τη πληροφόρηση και τη διαφάνεια, διότι περί αυτού πρόκειται. Ο Ασάντ δημοσιοποίησε πληροφορίε που ανησυχούν, ταράσουν, κυρίω για εγκλήματα πολέμου που διεπράχθησαν από τι ΗΠΑ. Παρά να λάβουμε υπόψη το έγκλημα, να λάβουμε υπόψη το έγκλημα, η κυβέρνηση θέλει να αποσιωπήσει, να σιωπήσουν οι φωνέ που ακούγονται. Θα πρέπει να ενταχθούμε σε αυτό. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τη δημοκρατία την ανοιχτή, τη διαφανή, ε, και να είναι υπεύθυνε οι πράξεις μας. Το θάρρος του είναι αυτό που κρίνεται σήμερα. Εάν δεχθούμε να εκδοθεί ο Ασάνς, θα εκδώσουμε αύριο όλους εκείνους που δημοσιεύουν πληροφορίες ευαίσθητες, δημοσιογράφους του Guardian, της Moon, του Spiegel, που δημοσίευσαν έγγραφα ε, που έχουν βρει από το Wikileaks. Η Γαλλία θα πρέπει να δώσει άσυλο στο Julian Assange και να υπερασπιστεί το χρώμα της διαφάνειας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, εκ μέρους του EFTD, το λόγο έχει ο William Dartmouth. Ευχαριστώ. Ας ξεκινήσουμε με μία πρόταση, μία αρχή. Δεν είναι καλή ιδέα οι πολιτικοί να προσπαθήσουν να παρέμβουν σε μία νομική διαδικασία. Αυτό πραγματικά είναι μία πολύ κακή ιδέα ο διαχωρισμός πολιτικής και νόμου είναι στο επίκεντρο των αξιών της δυτικής δημοκρατίας. Στην περίπτωση του κυρίου Τζούλιαν Ασάνς ε, συνελήφθη ε, προσήχθη στο δικαστήριο και καταδικάστηκε διότι θεωρήθηκε ότι ήταν ένοχος ε, παραβίασε τις συνθήκες εγγύησης. Είναι διαφορετικέ οι κατηγορίε του Χάκιν και άλλε παρεμφερεί κατηγορίε που τα παγκέθηκαν στι ΗΠΑ. Αυτέ είναι τα αντικείμενα τη ακρόση περί εκδόσεως. Η ακρόση θα λάβει χώρα ενώπιον δικαστού Βρετανού. Και αυτό που είπε το Συμβούλιο ήταν από τα γεγονότα ασφαλμένο. Ο Υπουργό Εσωτερικών δεν είναι αυτό που αποφασίζει. Πολλοί, εμού συμπεριλαμβανομένου, ε, διαφωνούσαν ε, με κάποιε αποφάσει δικαστών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά κανένα σοβαρό άνθρωπο αμφισβητεί την αντικειμενικότητα και τον επαγγελματισμό του αγγλικού δικαστικού κλάδου. Παρόλα αυτά, η κυρία Γκόμεζ και άλλοι συνάδελφοι θέλουν η νομική αυτή διαδικασία να υπόκειται σε πολιτική παρέμβαση. Αυτή είναι η τελευταία μου ομιλία στο Κοινοβούλιο και πρέπει να διαφωνήσω. Το να συζητάμε, να εξαρτούμε, να επηρεάζουμε πολιτικά τη δικαστική διαδικασία είναι κάτι που είναι αντίθετο όχι μόνο στις δυτικέ αξίες, αλλά κυρία Ζολή, εναντίον όλων των θεσμών της δημοκρατίας. Θα πρέπει εμείς ως πολιτικοί να αφήσουμε το θέμα, το νομικό θέμα του Τζούλιαν Assange στην ησυχία του, να μην το αγγίξουμε. Τώρα, ποιε ήταν οι αρχικέ νομικέ διαδικασίε που οδήγησαν στο να ξεφύγει, να παραβεί τι συνθήκε για την εγγύησή του, του κ. Σάντ. Ήταν το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη. Και αυτό το ένταλμα σύλληψη δεν εκδόθηκε από Σουηδό δικαστή, αλλά από Σουηδό εισαγγελέα. Παρά τα αυτά, με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, δεν υπάρχει πραγματική υπεράσπιση κατά της έκδοσης και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Ακούμε πολλά εδώ περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άρα το, οι σοσιαλιστές, οι φιλελεύθεροι, οι Βρετανοί φιλελεύθεροι, όλοι οι υποστηριχτές του ευρωπαϊκού υπερκράτους που δεν σκέφτονται καν, είναι οι ίδιοι άνθρωποι εκείνοι που είναι μεγάλοι υποστηρικτές του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Οι προσπάθειες που κατέβαλαν για την προστασία πολιτικών δικαιωμάτων και για το ευρωπαϊκό τέλμα σύλληψη είναι πολύ ασφαλμένε προσπάθειες, όπως και στην περίπτωση του κυρίου Σάνς. Η προσπάθεια που καταβάλατε για προστασία πολιτικής ελευθερίας και για σωστές νομικές διαδικασίες κολλάνε στο καλέ. Και όλα εν ονόματι μεγαλύτερης ολοκλήρωσης. Εάν αυτοί οι άνθρωποι σκεφτόταν, ξανασκεφτόταν. Σας εκλυπαρώ, σας παρακαλώ να το ξανασκεφτείτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριο Τέλειος Κούλογλου από την ΚΟΕ έχει το λόγο. Άκουσα δύο πόντιους πιλάτους ε, σήμερα. Είμαστε υπέρ ε, των καταγγελόντων, αλλά δεν έχουμε αρμοδιότητες. Το Συμβούλιο και η Κομισιόν. Εδώ πέρα όμως είμαστε εμείς πολιτικό σώμα. Μπορούμε να έχουμε μια πολιτική άποψη για τα γεγονότα. Ακούστε τι γίνεται. Ας υποθέσουμε ότι ένας Ευρωπαίος δημοσιογράφος γράφει κάτι ή κάνει μια αποκάλυψη ε, για το Ιράν. Εάν ο Ασάνς εκδοθεί, υπάρχει ένα προηγούμενο εδώ. Δηλαδή, το Ιράν θα μπορέσει